Διάφορε επιτροπές αποφάσισαν να αρχίσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 69C παράγραφος 1 του ε, κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εκθέσεις που ε, δίνουν την εντολή για τις διαπραγματεύσεις αυτές είναι ε, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 69C παράγραφος 2 Μέχρι αύριο ε, αριθμός μελών πολιτικών ομάδων μπορούν να ζητήσουν η απόφαση ε, να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις να τεθεί σε ψηφοφορία. Σε αντίθετη περίπτωση, μόλις εκπνεύσει αυτή η προθεσμία που είναι 5η 30 Νοεμβρίου στις 12